Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης διατίθενται. Είναι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις, λέει ο πρόεδρος. Αν όχι, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα.